Λοιπόν, στο θέμα της ψηφοφορίας. Πρόκειται για την ε, παράταση θητείας εξεταστικής επιτροπής. Το, η διάσκεψη των Προέδρων έχει προχωρήσει στη, στον έλεγχο όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές της κακοδιοίκησης ε, κατά την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και την ομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Η Επιτροπή Πάνα θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω εργασία και ότι όλες οι αποστολές, ε, διερευνητικές ε, αποστολές ε, για ειδικέ μελέτες είναι ακόμα απαραίτητοι. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν βάσει των μέχρι τώρα διερευνήσεων και όλες οι συμμετέχουσες πλευρές θεωρούν ότι η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να συνεχίσει την εργασία της έτσι ώστε να την ολοκληρώσει. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται και γίνεται δεκτή η παράδοση.